Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη συνεδρία της Επιτροπής μας. Καταρχήν, η έγκριση της ημερησίας διάταξης, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Έγκριση των πρακτικών 21 με 22 Δεκεμβρίου και πάλι εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Σημείο 3. Οι υπηρεσίες στους ε, λιμένες. Και δίνω το λόγο στην κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Ένα διαδικαστικό θέμα για την ψηφοφορία που θα κάνουμε σήμερα. Βάση του άρθρου 73. Γιατί προχωρούμε κατευθείαν στην απόφαση για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις. Λόγω του ιστορικού <clears throat> αυτού του θέματος και του ιστορικού της στην προηγούμενη θητεία. Ίσως το θέμα αυτό χρήζει περισσότερης εξέταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την εθνική ισορροπία στην ομάδα διαπραγμάτευσης και άλλους παράγοντες. Γιατί η ομάδα διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να λάβει υπόψη και την παρουσία ατόμων που δεν είναι απλώς σκιώδεις εισηγητές. Αν πάρουμε αυτή την απόφαση θα έπρεπε λογικά να πάει πρώτα στην Ολομέλεια, τουλάχιστον θα πρέπει να καθυστερήσει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σήμερα, θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση, αλλά η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αφαιθεί για μια μεταγενέστερη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέγει ο πρόεδρο. Το καταγράφουμε. Εντάξει, θα πάμε στην ψηφοφορία και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, κάνουμε καταρχήν ένα έλεγχο. Ψηφίζετε όπως θέλετε, ναι ή όχι, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Με μικρόφωνο θέλετε να παρέμβετε, παρακαλώ. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο σας. Διαδικαστικό. Ναι. Ο κύριος Τέιλορ λέει «Λόγω της πολιτικής ευαισθησίας του θέματος αυτού και το γεγονός ότι η Κομισιόν προσπαθεί να πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει για το θέμα αυτό τα τελευταία 11 χρόνια. Και επειδή υπάρχουν πολλές ε, απόψεις ε, στεναρές από τη μια ή από την άλλη πλευρά σε σχέση με το θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να εξασφαλίσει ότι είναι ισχυρή η εντολή του πρωτού προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Και αυτό αφορά και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γι' αυτό ζητούμε να υπάρξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια προτού γίνει η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Ήθελα λοιπόν να έχω τη θέση του εισηγητή για το θέμα. Ο εισηγητής δεν θέλει να λάβει το λόγο. Ας το αποφασίσει η Επιτροπή, λέει ο κ. Φλέκενστάιν, εκτός μικροφώνου. Εξαρτάται από την θέση της Επιτροπής, που ο εισηγητής. Εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Εντάξει, η δοκιμαστική ψηφοφορία λειτουργήσε σωστά. Περνάμε στην τροπολογία 99 ως 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 με 14 απορρίζεται. Τροπολογία 105 και 106. 105 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Πού είναι ο Πάουλ, πού είναι η Χάνα. Α, εδώ είναι. Ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. 26-18 δεκτή. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Εκπίπτει οι υπόλοιπε μέχρι τη συμβαστική 2. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία επαλήθευσης. Πέρας. 38-7. Καμία αποχή. Τέσσερα καλύτερα ψηφοφορία στη συμβαστική τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 356 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 356 άρχεται πέρας 20-24 απορρίπτεται 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 370 και 372 που είναι ταυτόσιμες. 374 λέει, 374 ναι, υπέρ. Ναι, 373, 372, 374 υπέρ, κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 376 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 702 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 704 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 705 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 706 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται έλεγχος έλεγχος 107 έλεγχος άρχεται πέρας 18.26. 26 απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Απόχειας απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Απόχειας έλεγχος. Για την 111 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Το διαπίστωσα, δεν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εντάξει. Τώρα είναι εντάξει. 21-23 απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για τη δύο άρχεται η ψηφοφορία πέρας 21-24 απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1-1-4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος καλά έλεγχος για την 114 άρχεται Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει. Τώρα εντάξει, 25-20 εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 115. Πάλι περισσεύει ένας. Από το έλεγχο. Μα δεν γίνεται τώρα αυτό να γίνεται συνέχεια. Κι άλλος ένας, κι άλλος ένας. Εντάξει, τώρα εντάξει. 22-22 απορρίπτεται. Ωραία, καλά το έλεγξαμε. Συμβαστική 18, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 19, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 20, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21, όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, τροπολογία 143. 143. Υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται την Με 143, <clears throat> άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου. Πέρας. Απερίφθη πράγματι. Συμβαστή 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστή 22. Όχι. Όχι. Τροπολογία 155. Και 156. Υπέρ. υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 179. Άρχεται. Πέρας. 22-23 απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος και για τη 17. Άρχεται. Πέρας. 23-22 εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 148 άρχεται πέρας 21-24 απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 190 πέρας 24-21 εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.19 υπέρ κατά αποχές <clears throat> έλεγχος για την 219 άρχεται Πέρας. 19-26 απορρίπτεται. 2-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 218. Άρχεται. Πέρας. 26-19 εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29-13 και μία αποχή εγκρίνεται. Περνάμε στο νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28-14 εγκρίνεται. Και τώρα η εντολή διαπραγματεύσεων. Πάλι μονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. 24-14 με 7 αποχές. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος.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 Επομένω δεν γίνεται δεκτή η εντολή διαπραγματεύσεων. Κάνουμε μία σύντομη διακοπή γιατί θα αργήσει λιγάκι ο κύριος Υπουργός. Ή η κυρία Υπουργός.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

I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, ίσως. So, nachdem wir eine Viertelstunde Pause Κάναμε λοιπόν το διαλυματάκι μας για ένα τέταρτο, αλλά μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μαζί μου δύο υπουργούς τον κύριο Φρανσουά Μπάου, ο οποίο είναι ο Υπουργό Ανάπτυξη και Μεταφορών του Λουξεμβούργου, και την κυρία Σούλφαν Χάχεν, η οποία είναι Υπουργό Μεταφορών Υποδομών στο, στην Ολλανδία και είναι λοιπόν μια πρεμιέρα για μας να έχουμε μαζί δύο υπουργούς. Σας ευχαριστώ και τους δύο που είσαστε εδώ παρόντες μαζί μας. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί την προηγούμενη και την τωρινή Προεδρία του Συμβουλίου. Ο κύριος Μπαου θα μιλήσει για τα πεπραγμένα της δικής τους Προεδρίας και η κυρία Φανχάχεν για τα σχέδια της Ολλανδικής Προεδρίας. Θα κάνουμε μια σύντομη παρέμβαση οι δύο Υπουργοί και μετά θα προχωρήσουμε σε μια κοινή συζήτηση. Και μετά φυσικά οι δύο Υπουργοί θα λάβουν τον λόγο. Κύριε Μπάους, ξεκινώ με εσάς. Euh, Ευχαριστώ πολύ, Μάικλ, για την ε, εισαγωγή αυτή και θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι νέο ότι εγώ ως εξερχόμενος υπουργός της προηγούμενης προεδρίας ε, βρίσκομαι ταυτόχρονα με την κύρια Σούλτς ε, εδώ για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα και αυτό που δεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ προεδριών μπορεί να λειτουργήσει. Λουξεμβουργενή Προεδρία είχε μια εξαιρετική συνεργασία με την ε, τρέχουσα Προεδρία, την Προεδρία τη Ολλανδίας. Είχαμε εξαιρετικές επαφές με την κυρία Σούλτς σε όλη τη διάρκεια τη δική μας προεδρία και μπορέσαμε να προετοιμάσουμε μαζί τα αντίστοιχα θέματα και τώρα Ω Λουξεμβούργοι συνεχίζουμε την παρακολούθηση των θεμάτων κατά την Ολλανδική Προεδρία, των θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε εμεί. Θέματα μάλιστα στα οποία σημειώσαμε κάποια επιτυχία. Όταν είχα έρθει την άλλη φορά πέρυσι στο Κοινοβούλιο για να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας, ε, είχα εκφράσει την πρόθεσή μου να μην εργαστούμε σε εκατοντάδες ε, θέματα, αλλά να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη ε, θέματα. Θέματα, δεν θέλω να πω ότι ήμασταν σίγουροι ότι θα καταφέρναμε καλά αποτελέσματα εκεί, αλλά που είχαν αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και επίτευξη αποτελεσμάτων να συζητήσουμε δηλαδή σε βάθος ορισμένα θέματα αντί να συζητάμε πολλά θέματα επιφανειακά χωρίς το τέλος να έχουμε κάποιες απτές, ε, ε, κάποια απτά επιτέγματα να καυχηθούμε. Ε, στην νομοθετική πτυχή επικεντρωθήκαμε στις δύο ευαίσθητες πολιτικά προτάσεις του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους. Θα ξεκινήσω από αυτό το θέμα λοιπόν. Είχα ε, παρευρεθεί τον Οκτώβριο εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου μετά από το Συμβούλιο της 8 Οκτωβρίου. Ζητά συγγνώμη ο κύριος Υπουργό. Ε, ήρθα λοιπόν εδώ στην Επιτροπή σας τον Οκτώβριο για έναν απολογισμό μετά από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται να μπω στις λεπτομέρειες τώρα, απλά να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαι ικανοποιημένος που επιτύχαμε το συμβιβασμό του 8 Οκτωβρίου. Και όπως σας είχα υποσχεθεί τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε αμέσως τους τριμερείς διαλόγους. Τρεις τέτοιοι διαλογοί έλαβαν χώρα στη δική μας Προεδρία μαζί με τους Ολλανδούς συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν δραστήρια σε αυτούς τους τριμερείς διαλόγους. πρόεδρος αναφέρει ότι χτυπάει το τηλέφωνο του κύριου Υπουργού. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αμέσω του τριμερεί διαλόγου, όπω είπα, μαζί με την ε, Ολλανδική Προεδρία, στη διάρκεια τη δική μα Προεδρία, ώστε να προετοιμάσουμε το φάκελο και να τον ολοκληρώσουμε το αργότερο το Μάρτιο, Απρίλιο φέτος του 2016. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω για τη δέσμευσή τους και τον επαγγελματισμό τους στη δική μου ομάδα αλλά και το σύνολο της γραμματείας, τις αντίστοιχες ε, νομικές υπηρεσίες ε, που επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο. Διαφορετικά δεν θα είχαμε καταφέρει να έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα. Ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για τι διαπραγματεύσει του τέταρτου πακέτου σιδηροδρόμων και εκεί η κοινή προσέγγιση των δύο διαδοχικών προεδριών αποδείχθηκε ωφέλιμη. Όπως σας είπα, σχεδιάσαμε μαζί ε, τα θέματα αυτά και έλαβαν χώρο όπως είπα, τριμερείς διάλογοι όπου ε, εξετάσαμε διάφορα ζητήματα, καταφέραμε να βρούμε κάποιες εξηγήσεις και να εξηγήσουμε τους διάφορους συμβιβασμούς και τις λύσεις και μέσα ως Κοινοβούλιο. Αυτά κάναμε κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Αυτή την εβδομάδα πρέπει να λάβουν χώρα ακόμη τρει τριμερεί διάλογοι όπου θα εξεταστούν πιο συγκεκριμένα σχέδια κειμένων. Όπω σα είχα εξηγήσει τον Οκτώβριο, σα είχα εξηγήσει τότε τι λεπτομέρειε του συμβιβασμού, οπότε δεν πρέπει να τι ξαναεξηγήσω σήμερα. Απλά να υπενθυμίσω ότι καταφέραμε τότε να επιτύχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Ε, ο συμβασμό που επιτεύχθηκε ήταν ιδιαίτερα εύθραυστο στις 8 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο του Συμβουλίου, όλα τα κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ ε, του κειμένου παρότι είχαν εκφράσει δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο είχε σχεδιαστεί το κείμενο όταν καθίσαμε στο τραπέζι. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι καταφέραμε να επιτύχουμε κάποια ισορροπία με όλες τις ε, τροπολογίες που κάναμε, με κίνδυνο φυσικά να χάσουμε την υποστήριξη διαφορών αντιπροσωπιών. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή την ισορροπία που ξεκινήσαμε εμεί θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε ώστε να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό μέσα στου επόμενου μήνε όπως έχουμε υποσχεθεί. Για να κλείσω θα ήθελα να επενέσω την επικοδομητική στάση των όσων συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει, του Κοινοβουλίου των εισηγητών χάρη στην οποία καταφέραμε να βρούμε λύσεις για θέματα επί της ουσίας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς πρέπει να λειτουργεί, πιστεύω, η συναπόφαση. Να συνενώνουμε τις δυνάμεις μας αντί να καταλήγουμε σε παράλυση. Ε, με χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερα όλο αυτό που επιτύχαμε. Το Συμβούλιο, ξέρετε, εκφύσεως ε, πρέπει να είναι πιο ρεαλιστικό όσον αφορά τις αποφάσεις του. Έχουμε πολύ μικρότερο περιθώριο λιγμών σε επίπεδο Συμβουλίου. Ενώ το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, προσφέρει περισσότερες διαφορετικές απόψεις, μια διαφορετική προοπτική και πιστεύω ότι συνδυάζοντας αυτές τις δύο προσεγγίσεις θα καταφέρουμε να δώσουμε την οριστική του μορφή σε αυτό το κείμενο. Η εσωτερική ναυσιπλοεία τώρα η Λουξεμβουριανή Προεδρία ξεκίνησε τη διαπραγματεύση για την πρόταση οδηγίας σε σχέση με ε, τις τεχνικές προδιαγραφές για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Δεν έχει ακόμα ε, υπάρξει κάποια συμβαστική λύση, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν οι Ολλανδοί συνάδελφοι και τώρα έρχεται το εκανθόδε ζήτημα της ε, αεροπλοείας. Όπως εξήγησα τον Ιούλιο πέρυσι, στον τομέα αυτό τα προσκόμματα στις εργασίες δεν έχουν αλλάξει. Δυστυχώς λόγω της πολιτικής κατάστασης που γνωρίζετε όλοι ε, τα πράγματα δεν πρόκειται να ξεμπλοκώρουν τόσο γρήγορα. Όπως είπα πριν από 6 μήνες ε, συμμερίζομαι την άποψη ότι ο νομοθετής πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του σε αυτό τον τομέα και ειδικότερα όσον αφορά την πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο εμείς υιοθετήσαμε αυτό το φάκελο στην Κορεπέρ και συζητήσαμε με την Κομισιόν για την αναγκαιότητα αναθεώρησης των σημερινών κανονισμών. Ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, με χαροποιείται ότι η Κομισιόν παρουσίασε τη στρατηγική της ε, στρατηγική για την αεροπορία στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και αυτό θα επανεκκινήσει, ελπίζω, τη συζήτηση και ελπίζω ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι Ολλανδοί συνάδελφοι θα καταφέρουν ε, να φτάσουν στην τελική φάση σε ορισμένα θέματα. Τώρα, ένα νομοθετικό θέμα που πρότεινα εγώ με δική μου πρωτοβουλία ε, στο πλαίσιο συζητήσεων προς Ανατολισμού, όπως είχαμε πει στην αρχή της Προεδρίας μας, ε, θα κάναμε δύο συζητήσεις προς Ανατολισμού στο Συμβούλιο, ώστε να δώσουμε δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν το όραμά τους στην Κομισιόν. Αυτό φυσικά είναι σημαντικό διότι όπως γνωρίζουμε όλοι οι Κομισιόν ε, ε, εργάζεται σε αυτούς τους φακέλους και με αυτόν τον τρόπο εμείς θέλαμε να επηρεάσουμε τις εργασίες της Κομισιόν μέσω των συζητήσεων του Συμβουλίου. Αρχικά λοιπόν στον Οκτώβριο βάσει των κατευθύντηρων γραμμών για την πολιτική μεταφορών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βαζόμενη στη Λευκή Βίβλο και στην εκθέση του κ. Βαντεκάμπ ε, το Δεκέμβριο εξετάσαμε τις ε, κοινωνικές πτυχές των οδικών μεταφορών. Θέλησα εγώ να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα πριν ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν ε, σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Οι ανταλλαγές μας πιστεύω ήταν ειλικρινείς και ωφέλιμες, κυρίως για την Κομισιόν, διότι η Κομισιόν ε, είδε πλέον ποιες είναι οι τάσεις συγκεκριμένα στα κράτη-μέλη. Δεν ξεχνάμε φυσικά την οδική ασφάλεια, η οποία δεν πάβει να αποτελεί προτεραιότητα της κοινή μας δράσης. Ε, ανταλλάξαμε πολύ ειλικρινά απόψεις για τις καλύτερες πρακτικές με την Κομισιόν και αναφερθήκαμε και στο δίπλωμα οδήγησης ε, ε, με σύστημα πόντων για, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ατυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς είναι ένα φλέγον θέμα στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο επισταμένα. Επίσης οργανώσαμε ένα άτυπο συμβούλιο. Ε, πρώτη φορά οργανώθηκε ένα συμβούλιο που εξέτασε τους ίδιους τρόπους ε, μεταφορών όπως το ποδήλατο και αναφέρθηκε και στην πρόθεση των λιγότερο ρηπενών τρόπων μεταφοράς. Ε, σε μια λοιπόν άτυπη συνάντηση αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα μέσα μεταφορών ε, η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη, μεγάλη προσέλευση και σε υπουργικό μάλιστα επίπεδο και χαίρομαι ιδιαίτερα που και η δική σας Προεδρία και ο Προεδρός σας ε, ε, ήταν μαζί μας και εξέφρασε την υποστήριξή του για τους τρόπους αυτούς μεταφοράς. Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του ποδηλάτου και για τις κοινωνικές και οικονομικές τυχές του και οι Υπουργοί Μεταφορών υιοθέτησαν ένα ψήφισμα για το ποδήλατο ως τρόπο μεταφοράς, ως μέσο μεταφοράς και η δήλωση αυτή, η διακήρυξη αυτή επικυρώθηκε στο επίσημο Συμβούλιο 8 Οκτωβρίου από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης και τώρα ένα αποκτήστη μισιό να λάβει υπόψη το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης. Το ποδήλατο φυσικά δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά μπορεί να συμβάλλει στην επίλυσή τους. Και εγώ θα συνεχίσω να προωθώ το θέμα αυτό, όπω έκανα ανέκαθεν. Αυτό είναι ένα σύντομος απολογισμός Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Είμαι τώρα στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω στι προτάσει, τι επικρίσεις, τι ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ και για τη συμβολή σα ε, και τι προτάσει σας κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας και τον απολογισμό που μας παρουσιάσετε και δίνω τώρα το λόγο στην Ολλανδική Προεδρία. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Μάικλ, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών, με μεγάλη μου τιμή σα δίνω το λόγο σήμερα ω πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών και προβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια τη Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου και αναμφίβολα η συνεργασία, κατά τη γνώμη μου, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Ε, Κάποιου του έχω συναντήσει και στο παρελθόν, ελπίζω να γνωρίσω και τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών ε, μέσα στα επόμενα εξάμεινα. η συνάντηση του Δεκεμβρίου, σε εκείνη τη συνάντηση, χρησιμοποίησα την εικόνα ενός ε, διθέσιου ποδηλάτου για να απεικονίσω και την ε, συνεργασία μου με τον Φρανσά ε, Μπάους. Την Προεδρία του Λουξεμβούργου, ήταν τότε η Λουξεμβουργική Προεδρία στο τιμόνι και εμείς η Ολλανδική Αντιπροσωπεία στην πίσω θέση, ετοιμαζόμενοι να πάρουμε και εμείς το τιμόνι. Σήμερα είναι και οι δύο υπουργοί εδώ που είναι και μια κάτι το καινοτόμο, κάτι το καινούργιο Και ο Φρανσουά ήταν πολύ καλός συνοδηγό Στο κοινό μα ποδήλατο τώρα ήρθε η σειρά να πάρω εγώ το πιδάλιο. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι εταίροι μα, ε, Σλοβακία και Μάλτα, του Τρίου Προεδρία, ετοιμάζονται και αυτοί να πάρουν ε, την Προεδρία στο μέλλον. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ε, κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα και ελπίζουμε κιόλα να ανεβάσουμε ταχύτητα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πριν ε, περάσω σε συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα πρώτα να σα ε, αποστείλω ένα γενικό μήνυμα ω Προεδρία του Συμβουλίου. Πρώτα, χρειαζόμαστε μια συνεργασία για να έχουμε αυτά αποτελέσματα, να επικεντρωθούμε στα κέρια ζητήματα, στα οποία πράγματι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Άλλα ζητήματα μπορούμε καλύτερα να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δεύτερον, πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η καινοτομία. Και αυτό υπό δύο έννοιες. Η καινοτομία ως κινητής μοχλός για την βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, ενίσχυση της συνταγωνιστικής ισχύω τη Ευρώπης και η καινοτομία ε, ω ε, τρόπο ε, λειτουργία από πλευρά νομοθετικού πλαισίου και κανονιστικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευφυή e e και ε, λειτουργική προσέγγιση και για τις επιχειρήσεις, για τις startups, να ενισχύσουμε την δημιουργικότητα, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Μετά, σε ένα διοργανικό επίπεδο, θα πρέπει να επενδύσουμε σε μια καλή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Κομισιών και Συμβουλίου. Για την συνεργασία αυτή ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή για την Ευρώπη. Χρειάζεται μόνο να αναφερθώ στην ε, προσφυγική κρίση, στο, στη δρομοκρατία και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και βεβαίως ε, και τα σύνορά μας και το πώς αυτά επηρεάζουν ε, και τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγκυται μόνο στο κανονιστικό πλαίσιο και πάλι χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων και ενωμένοι να αναλάβουμε δράση. Δεν είναι μόνο η καλή νομοθεσία, αλλά και καλή εφαρμογή της νομοθεσίας. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο. Τώρα για την καινοτομία ανέφερα και την καινοτομία πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες για να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, γιατί βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας νέας επαναστατικής ε, βιομηχανικής επανάστασης και στον τομέα των μεταφορών θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα δούμε περισσότερες αλλαγές από ότι τον τελευταίο αιώνα. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα ενισχύοντας και προωθώντας ε, ευφυείς λύσεις σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και τις υποδομές. Ε, και έτσι νομίζω ότι θα έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, ε, λιγότερα τροχέα στους δρόμους και γενικότερα καλύτερη λειτουργία του, του συστήματός μας μεταφορών με μεγάλη έμφαση όμως ε, στην αυτόματη οδήγηση και στην διασυνδεδεμένη οδήγηση. Θα κάνουμε και ένα άτυπο συμβούλιο των, μεταφορών, ε, των Υπουργών Μεταφορών στο Άμστερνταμ μαζί με τον συνάδελφο Τζέρα Ντάσμαν και εκεί θα προσκαλέσουμε τους συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για ζητήματα μεταφορών και περιβάλλοντος για να διαρευνήσουμε μελλοντικές λύσεις για την βιώσιμη κινητικότητα. Και βεβαίως ε, καλό θα ήταν υπάρχει και αντιπροσωπεία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συμβάλλει σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν να σας δω όλους εκεί. Και τρίτον, έχουμε τις ε, καλές ε, σχέσεις συνεργασίας. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυτές οι καλές σχέσεις. Θέλουμε να, να είμαστε δίκοι, διαφανείς και αποτελεσματικοί. Ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί σωστά παρόλες τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουμε. Και έχουμε θέσει κάποιες βασικές προτεραιότητε όπως είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ισχύ ε, της ε, βιομηχανίας ε, αεροπλοείας μας στην Ευρώπη. Και την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο Σχίπχολ είχαμε μια συνάντηση, άτυπη συνάντηση πολλών και υπουργών αλλά και διευθυντών εταιριών αεροπορικών εταιριών και τον Ιούνιο όμως θα γίνει μία αντίστοιχη συνάντηση όπου θα εξετάσουμε το λεγόμενο T-Days βεβαίω σε στενή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διατηρούμε λοιπόν ε, τι ε, καλέ σχέσει συνεργασία. Ε, για να γίνει αυτό όμω πρέπει να επενδύσουμε και σε έναν αυτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω μέσα στι επόμενου μήνε να έχουμε καλά και θετικά αποτελέσματα σε στενή συνεργασία μαζί σα. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στου εξή φακέλου. Πρώτον, αεροπλοεία. Η στρατηγική της Κομισιόν ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης ε, στην Ευρωπαϊκή Συνόδο Κορυφής για την Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάικελ Βίμ, Χεσίν, Ντέρι Τρεματές. Ήταν μεγάλη μου χαρά να σας υποδεχθώ εκεί. Η Σύνοδος Κορυφής δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή αεροπλοεία είναι κέρια σημασία για τις οικονομίες μας, για την απασχόληση, την συνδεσιμότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε περιφερειακό και τοπικό και για την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Λάβουμε λοιπόν σαφή μηνύματα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκής αεροπλοεία και μάλιστα αυτό να αποτελέσει προτεραιότητα. Ε, βλέπω ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί πρόοδος ό,τι αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και τον ΣΕΖΑΡ και μάλιστα με έμφαση στην καλύτερη εφαρμογή τους. Η, Προεδρία, μάλλον ε, βλέπει ότι υπάρχει στήριξη για να προχωρήσουμε και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και ε, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και στον ΕΑΣΑ. Ε, υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις και σε ό,τι αφορά τις ε, εντολές διαπραγμάτευση, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κράτη του κόλπου, την, τις χώρες Asian και την Τουρκία. Όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούν και να βρουν κοινό έδαφο σε πολλού τομεί μέσα από επόμενου μήνε. Όπω για παράδειγμα στα σιδηροδρομικά. Στόχο είναι να υπάρξει συμφωνία ε, κατά προτίμηση πριν από το Πάσχα σε ό,τι αφορά το τέταρτο ε, πακέτο, να αξιοποιήσουμε την θετική δυναμική και είμαι σίγουρη ότι μπορεί να σημειωθεί επιτυχία. Όμως, Υπάρχουν κόκκινε γραμμέ, όπω είπε και ο Φρανσουά. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων και υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, την οποία δεν θα πρέπει να χάσουμε με τα κρατημέλη. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ευελιξία. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία, έχουμε την ίδια φιλοδοξία για την πρόταση για τι τεχνικέ προδιαγραφέ για τα σκάφη εσωτερική ναυσιπλοεία. Όπω ε, και στο πακέτο για τα συνδρομικά. ο προκάτοχο μου, Φανσουά Μπάου έκανε μια εξαιρετική δουλειά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μα για να βρούμε μια πρακτική λύση για να υιοθετηθεί η οδηγία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εναρμονισμένο τεχνικό καθεστώ σε όλη την Ευρώπη γιατί είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα και για μένα προσωπικά η ενίσχυση ε, της αυστερικής ναυσιπλογίας στην Ευρώπη. Για τους λιμένες, νομίζω ότι υπήρξε, ήμουν μάλλον διατεθειμένη να πω ότι υπήρξε καλή διαπραγμάτευση και θετική ψήφο για την εντολή σήμερα, αλλά δυστυχώ άκουσα ότι δεν επετεύχθη κάτι τέτοιο σήμερα το απόγευμα. Επομένω, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα πραγματική συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Ελπίζω όμω να ψηφίσετε και να υιοθετήσετε μία εντολή διαπραγμάτευση σύντομα και γνωρίζω ότι δεν έχω θίξει όλα τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η δική σας Επιτροπή. Ήθελα να θέσω κάποιες προτεραιότητες. Βεβαίως, με τις ερωτήσεις σας μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια επιπλέον ζητήματα. Κλείνοντας, ε, δύο λόγια για τον τουρισμό, παρότι δεν είμαι αρμόδια για αυτό το ζήτημα. Ο συνάδελφός μου, κ. Δεκάμπ, που είναι ε, προσκεκλημένος ε, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, είναι αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα, αλλά Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Για μας ε, η ανάδυση νέων ε, επιχειρηματικών μοντέλων σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και την ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα. Πρέπει να ενισχύσουμε την ποιότητα των ε, υπηρεσιών, των δεξιοτήτων, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά και μία εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά που είναι όλα αυτά απαραίτητες προϋποθέσεις για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό. Τέλος κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησα αυτή την εικόνα ότι το Λουξεμβούργο και οι κάτω χώρε οδηγούν ένα διθέσιο ποδήλατο. Όμως ε, Μάλλον καλύτερα σήμερα είναι να πούμε ότι οδηγούμε ένα τριθέσιο ε, ποδήλατο, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ε, που τραβήχτηκε στο Συμβούλιο Μεταφορών, στο οποίο μας προσκάλεσε ο Φανσφά. Νομίζω ότι από κοινού θα πρέπει να εργαστούμε, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν και θεωρώ ότι ε, και είναι και ο ρόλος μου να εκπροσωπήσω όλα τα κρατημέλη όσο μπορώ καλύτερα και να συνεργαστώ μαζί σας για ένα βιώσιμο μέλλον με απασχόληση, ανάπτυξη, ειρήνη και ευημερία και ε, δημόσια στήριξη για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο γύρο των συν... συντονιστών με τον κύριο Φαντελκάμπ πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και από πλευράς μου βεβαίω να καλωσορίσω και του δύο υπουργού. Θα ήθελα να απευθυνθώ πρώτα στον κύριο Μπάους και μετά στην κυρία Σουλς. Βεβαίως ε, είναι και ε, συνδέονται μεταξύ τους ε, και τα χαρτοφυλακιά τους, αλλά θα ήθελα να τα εξετάσω ξεχωριστά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ε, που έχουμε αυτή την, το νέο κόνσεπτ των δύο υπουργών. Γιατί είχαμε κάποιες εμφιβολίες ε, και με, για το Συμβούλιο, κατά πόσο όλα αυτά συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, αλλά ε, αυτοί οι δύο έχουν το πλεονέκτημα ότι γνωρίζονται καλά και από την Πενελούξ, αλλά ελπίζω αυτό να ισχύσει και για τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πείραμα αυτό. Θα δούμε όμως. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπάους για τα όσα μας είπε και για τις προσπάθειες που κατέβαλε, αλλά και για τα αποτελέσματα που επέτυχε. Πρέπει, όχι επειδή είναι και ο κύριος Ζουβάης εδώ συγκεκριμένα, αλλά πρέπει ρητός ε, να ευχαριστήσουμε και το επιτελείο των ε, Υπουργών, γιατί νομίζω ότι όλα πήγαν πολύ καλά. Ε, αναφερθήκατε στο συνδεδομικό πακέτο και η κυρία Σούλς το ανέφερε. Υπάρχει καλό κλίμα στο Κοινοβούλιο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μέχρι το Πάσχα να επιτευχθεί συμφωνία. Και με τη γενική προσέγγιση στις 8 Οκτωβρίου, νομίζω ότι κάνατε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για το να είδες, είναι σαφές ότι προχωρούμε και με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Για να είμαι ειλικρινή, Πρόεδρε, πάντα είμαι λίγο επιφυλακτικός ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική και τα ποδήλατα. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σας χόμπι, αλλά εμείς ε, στι κάτω χώρε έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά και στο ΕΛΚ ε, ευρύτερα, γιατί η επικουρικότητα είναι το παν. Και αν κάποιος ε, θέλει να κάνει μια ωραία πράσινη φιέστα, εντάξει, αλλά Ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τα ποδήλατα και την αστική κινητικότητα έχουμε και καλά παραδείγματα επί τούτου στην Ολλανδία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε. Αλλά όχι στην, ε, από πλευρά πολιτική, αλλά από πλευράς βέλτιστων πρακτικών. Πρόεδρε, έχουμε τρία χαρτοφυλάκια τα οποία συνδέουν τον κύριο Μπάου με την κυρία Σούλτ. Πρώτον, έχουμε το σκάνδαλο με τι εκπομπέ. Κανένα από του δύο δεν το ανέφερε. Ε, η COP21 είναι ένα θέμα που έθιξε ο κύριος Μπάους, αλλά το σκάνδαλο για τις εκπομπές ήταν πολύ σημαντικό θέμα και στην COP21. Το δεύτερο, το οποίο ανέφεραν και οι δύο υπουργοί, είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε το παλιό πακέτο για την αεροπλοεία. Ο κύριος Ανμπάχ ε, σίγουρα θα το αναφέρει. Ελπίζω φέτος

Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση ήταν μεγάλη επιτυχία με πολλές άτυπες συζητήσεις και από πλευρά της βιομηχανίας και βλέπω ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην καινοτομία. Η Ευρώπη εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καινοτομία. Εντάξει, να παράγουμε και ε, ατσάλι και μέταλλο, αλλά όχι και τόσο πολύ πια. η καινοτομία είναι αυτό που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για μας. Και χαίρομαι που μιλήσατε και για την εφαρμογή, γιατί θεσμοθετούμε τόνους νομοθεσίας, αλλά τελικά τίποτα δεν εφαρμόζεται. Και θα ήταν πολύ καλό, ε, κάτι το οποίο απασχολεί βεβαίως εσωτερικά την Ολλανδία, να υπάρξει ένα εσωτερικό ψηφιακό έγγραφο για τους ε, οδηγούς. Τώρα, ο κύριος Κράμερ, έχουμε και το δεύτερο αγαπημένο του χόμπι μετά τα ποδήλατα, που είναι ε, τα οχήματα, αυτόματης, τα αυτόματα οχήματα. Θα προχωρήσουμε και εκεί. Κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι επενδύσεις ε, στους μικρούς ε, δρόμους. Γιατί πολλά είναι τα κονδύλια που απευθύνονται στα TNT, όλα αυτά πολύ καλά εφαρμόζονται. Εντάξει, λίγο καθυστερούμε με τις άδειε, αλλά και σε σχέση με τη Γαλλία θα πρέπει, θα πρέπει να εξετάσουμε την μικρή ε, ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Μπάους, αγαπητή κυρία Σούλτς, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστώ και την διεύθυνση της Επιτροπής μας που έχει φέρει από κοινού τους δύο υπουργούς. Αυτό είναι μια πολύ καλή εικόνα. Ξεκινώ με αυτά που είπε ο κύριος Μπάους και τον ευχαριστώ καταρχήν για, τα, για την εξάμεινη προεδρία του Λουξεμβούργου. Είναι πράγματι αξιέπαινα αυτά τα οποία έκανε και οι προσπάθειες τους για το τέταρτο πακέτο σιδηροδρομικών θεμάτων. Να θέσω τώρα κάποια ερωτήματα σε εσά κύριε Μπάους ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη για τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με αυτό το πακέτο το τελευταίο εξάμεινο και πώς επίσης βλέπετε την ε, τεχνική πτυχή για τα θέματα αυτά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για το θέμα αυτό Περιμένουμε όμως να έχουμε την ε, άποψη του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω με ποιο τρόπο εσείς προβλέπετε να υπάρξει μια συμφωνία στον ε, Τρίλογο και πώς μπορείτε να συμβάλλετε σε κάτι τέτοιο. Έρχομαι τώρα στην κυρία Σούλτ Φανχάγεν. Κυρία Υπουργέ, αναφέρατε πολλά σημεία που είναι σημαντικά και θετικά για μένα για την Ολλανδική Προεδρία να σταθώ πρώτα με ένα θέμα που είναι κάπως ε, αμφιλεγόμενο και το οποίο έχετε περιλάβει στο πρόγραμμα σας ε, της Προεδρίας, λέτε ότι θα θέλετε να προωθήσετε με αποτελεσματικό τρόπο τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ. Ξέρετε όμως πόσο δύσκολος είναι αυτός ο φάκελος και ιδίω στη δική μου πατρίδα στη Γερμανία υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ποιες είναι οι δικές σας προσωπικές απόψεις για τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η Συμφωνία TTIP στον ευρωπαϊκό μεταφορικό χώρο, δηλαδή και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στον κατάλογο προτεραιοτήτων σας επίσης που διάβασα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα βέβαια, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό που λέτε για, τον, για τις οδικές μεταφορές. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι σας σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα και επίσης θα με ενδιαφέρει δική σας άποψη για το πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε την κοινωνική διάσταση στον ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών, δηλαδή συνδίκες εργασίας, ασφάλιση, αποδοχές των εργαζομένων στον τομέα αυτό, τι ρόλο θα πρέπει να παίξουν όλα αυτά και ένα τελευταίο σημείο <clears throat> και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερα γιατί έχετε ενδιαφερθεί για το θέμα των αυτονόμων οχημάτων, χωρίς οδηγό δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μαζί με άλλους συναδέλφους έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε το θέμα αυτό τόσο πολύ ώστε και η Κομισιόν θα έρθει να μας παρουσιάσει την άποψή της μετά από προφορική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της Ολλανδικής Προεδρίας για το θέμα αυτό και κατά πόσο συμφωνείτε και εσείς ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ταχύτερων Δυνατών θα πρέπει να μας παρουσιάσει μια πράσινη βίβλο για το θέμα των αυτονόμων οχημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Υπουργό και την κυρία Υπουργό εδώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πόσο καλά αυτό το διπλό ποδήλατο λειτουργεί. Μια χαρά με αυτές τις δύο πρόεδρες του Λουξεμβούργου και των κατοχωρών. Σας παρακαλώ να μην ξεχνάτε και την επόμενη Προεδρία της Σλοβακίας. Ε, εντάξει δεν λέω να εργαστούν ως τρόικα αλλά να αποτελέσουν μια ικανή συνέχεια του δικού σας ε, πολύ επιτυχημένου έργου. Τώρα, όσον αφορά το η τέταρτη δεσμε μέτρο για του σιδηροδρόμου, η πρόοδο που σημειώθηκε ήταν εξαιρετική κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Φυσικά το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί ίσω να μην είναι ακόμα το τέλειο, αλλά πιστεύω ότι θα ε, σημειώσουμε επιτυχίες της διαπραγματεύσεις και ότι θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες ε, του τεχνικού πυλώνα και του πολιτικού πυλώνα και ότι θα συμφωνήσουμε επί των κόκκινων γραμμών, διότι για παράδειγμα όσον αφορά τους ελέγχους κράτους λιμένα έχουμε πολλά κόκκινες γραμμές ε, για, σε αυτόν τον τομέα Ας δούμε πώς θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με τον κανονισμό για τους λιμένες. Αναφέρατε την ανάπτυξη των τεχνολογικών πληροφορικής και τις καινοτομίες. Θα ήθελα να εκφράσω κάποια ανησυχία για τους τομείς αυτούς. Όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση και το δομέα των μεταφορών, γνωρίζουμε ότι η Προεδρία των Κατοχωρών θα επιδιώξει λύσεις Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των διαφορών χωρών. Το σύστημα Σέγγεν αυτή τη στιγμή διατρέχει κίνδυνο. Και αυτό επηρεάζει την κατάσταση της μεταφορές με αρκετό κόστος. Για παράδειγμα η γέφυρα Ερεσούντου που συνδέει την Δανία και τη Σουηδία πλέον έχει ελέγχους πάνω στο δρόμο και μπλόκα στους δρόμους ε, και έτσι οι μεταφορές εκεί αρχίζουν να κοστίζουν πολλά. Υπάρχει κίνδυνος ισχυρού πλήγματος τελικά στον τομέα των μεταφορών όλα αυτά. Όλες αυτές οι σοβαρές συνέπειες πρέπει να τις λάβουμε στα σοβαρά. Όταν προγραμματίζουμε το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη και τους οικονομικούς πόρους που σχετίζονται με αυτό, όλα αυτά αφορούσαν διασυνοριακά έργα. Αν τώρα ασκούμε πολιτική πίεση για να προχωρήσουν αυτά τα έργα, και βρεθούμε σε ένα χώρο Σέγγεν ε, που ξαφνικά αποκτά ξανά σύνορα θα χάσουμε χρήματα σε αυτά τα διασυνοριακά έργα. Απλά διότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα αρχίσουν να υπάρχουν ξανά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις απόψεις κύριε ε, Υπουργέ. Τι είδους λύσεις μπορούμε να αναμένουμε. Ευχαριστώ και Μάιστερ. Έχει Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο υπουργούς. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ καλό που ο Ρόμπερτ Σίλε αναφέρθηκε στην δύσκολη κατάσταση που γενικά αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Νομίζω και οι δύο προεδρίες, και η Λουξεμβουργική και η Ολλανδική, έχετε αναλάβει την ε, προεδρία σε μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε πολλές φορές σε σχέση με την πολιτική μεταφορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κλείσουν πάλι τα σύνορα, πώς θα εξασφαλίσουμε να έχουμε παραγωγός πρακτικές όπως ολοκληρωμένη έκδοση εισιτήριων στο συνδρομικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. του Λουξεμβούργου. έχει κάνει ό,τι μπορεί για να τα πετύχει αυτά τα πράγματα. Θέλω να ευχηθώ και στην Ολλανδική Προεδρία και εσείς να καταφέρετε να φέρετε τις σωστές ε, αποφάσεις ανεξάρτητα από τα θέματα των μεταφορών που να εξασφαλίσουν την διατήρηση της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Αυτό είναι η γενικότερη προτεραιότητα. Και τώρα αναφερόμενοι στην Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών. Φυσικά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα το Λουξεμβούργο για το τέταρτο συνδεδομικό πακέτο και οι κάτω έχουν παρακολουθήσει όλες αυτές τις θετικές συμφωνίες και βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πρόοδο. Βέβαια, όταν γίνεται η διαπραγματεύση μόνο σε επίπεδο εμπειρογνώμων, δεν είναι κατά ανάγκη καλύτερα τα πράγματα. Το θέμα της, ε, των ε, λιμένων, βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα το, το Λουξεμβούργο. Για την ε, αεροπλοεία, ξέρουμε ότι υπάρχει εμπόδιο σε μια συμφωνία και είχε ένα πλεονέκτημα το Λουξεμβούργο, μια μικρή χώρα με μεγάλη διπλωματική ικανότητα θα μπορούσε ίσω να επιτύχει περισσότερα πράγματα έναντι των μεγάλων χωρών και τώρα φυσικά είναι η σειρά της, ε, των ε, Ολλανδών σε ό,τι αφορά τους ενίου ευρωπαϊκούς εθέρες και τα δικαιώματα των επιβατών να μπορέσει να προχωρήσει τα θέματα αυτά. Και τώρα στρέφουμε σε εσά, ε, κυρία Φανχάγεν. Να μην τίθεται πλέον ένα θέμα κυριαρχικότητα στους εθέρες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα την κινητικότητα των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει λοιπόν για ορισμένους τέτοιους λόγους ε, υποτιθέμενης ε, κυριαρχικότητας και τέτοιων προβλημάτων τα πράγματα να μείνουν παγωμένα. Είδαμε τι έγινε στην COP21 στο Παρίσι, που όλοι έχουμε υπογράψει αυτή τη συμφωνία, γιατί ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε λιγάκι την κατάσταση του κλίματος στον πλανήτη μας και εκεί λόγω μερικών λεπτομεριών υπήρξαν εμπόδια να υπάρξει και μια συμπερίληψη του τομέα της αεροπορίας, κάτι που θα έχει μεγάλη σημασία για τις εκπομπές. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί και θα ξεπεραστεί. Το ποδήλατο, ναι βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνατε μια διάσκεψη για την ποδηλασία, βλέπω τον πρόεδρό μας να χαίρεται ιδιαίτερα και αυτό φυσικά είναι κάτι που ταιριάζει όχι μόνο στο Λουξεμβούργο αλλά κυρίως στην Ολλανδία η κίνηση με ποδήλατο. Και επομένω είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ την, ε, τις μεταφορές στις πόλεις, βέβαια στον τομέα της υπαίθρου είναι λιγότερο σημαντικό. Και πάλι για την Ολλανδική Προεδρία μιλήσατε για τα θέματα της καινοτομίας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα τη καινοτομία, γενικά για όλε τι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και στον τομέα τη ασφάλεια των μεταφορών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λένε πολλοί ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει μόνο του αυτόνομα, χωρί οδηγό, ένα γιοταχή ή ένα φορτηγό μπορεί να είναι πολύ πιο ασφαλέ από ένα με οδηγό. Βέβαια, είναι σημαντικό να δούμε κατά ποιε προποθέσει μπορεί να γίνει αυτό και περιμένω να αντιμετώπισει και η δική σα Προεδρία το θέμα και τη αλυσίδα μεταφορών και ε, παραδόσεων προϊόντων που μπορεί να βοηθηθεί πολύ περισσότερο με την ψηφιοποίηση και να έχουμε μια πρόθεση της λεγόμενης smart mobility οπότε να μειώσουμε το άχθος των μεταφορών. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα ε, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά για το τέντι να δώσετε την απαραίτητη έμφαση, αλλά θα ήθελα να διατηρήσουμε αυτή την εικόνα που έχουμε για τους ε, διάβλους στην Ευρώπη. Αυτό είναι εμβληματικό μιας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης ενός προβλήματος όπως είναι οι μεταφορές για τα λιμάνια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν πέρασε εύκολα η απόφαση ε, στο, στην Επιτροπή μας προηγουμένω, είπατε ότι δεν υπάρχει πολύ περιθώριο λιγμών. Ελπίζω ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Συμβουλίου θα υπάρχει και κάποιο μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών. Και τέλος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον συναδελφό μου, το θέμα της TTIP. Και εγώ θα ήθελα να δω να προχωράει αυτή η συνεργασία. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε πλεονεκτήματα στην Ευρώπη αλλά είμαι και σκεπτικιστική γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις ΗΠΑ εναντί της Ευρώπης και θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε στον τομέα αυτό και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Μάια Κίλενεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους υπουργούς. Μου αρέσουν τα όσα λέτε, ε, ε, ε, βαγόνια, διασύνδεση μεταξύ τους, νέα βαγόνια. Ελπίζω όλες αυτές οι πρακτικές να περάσουν και στις επόμενες προεδρίες ως ιδέες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λουξεμβούργο για την επιτυχή του Προεδρία και εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Ολλανδική Προεδρία. Έχω μια ερώτηση για το Λουξεμβούργο και μια για τις κατοχώρες. Πρώτα προς το Λουξεμβούργο, προς την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Τι είδου κληροδότημα πιστεύετε ότι αφήνεται στην επόμενη Προεδρία όσον αφορά το, την τέταρτη δισμή μετρών για τους σιδηροδρόμους. Τι προκλήσεις πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσουμε ε, μελλοντικά για να καταφέρουμε να επιτύχουμε μία λύση μέχρι το Πάσχα. Για τις κάτω χώρες τώρα μια ερώτηση. Οι διάφορες υπηρεσίες για ε, πληροφορικής και το ψηφιακό θεματολόγιο πώς θα βελτιώσετε την νομοθεσία. Ε, για να βοηθήσετε τις νέες επιχειρήσεις, τους νέους επιχειρηματίες ε, για να δημιουργηθούν ευκαιρίες πώς πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να φέρετε τα δικαιώματά τους ε, και ε, τα ωφέλη τους στο ίδιο επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω βάλει και εγώ τον ε, εαυτό μου στον κατάλογο από τη δική μου πολιτική ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές μας και εύχομαι να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάους για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και ελπίζω ότι και η Προεδρία των κάτω χρόνων θα συνεχίσει αυτή η θαυμασία συνεργασία. Αναφέρθηκε πάρα πολύ εδώ ο δικός χάρτης για τα ποδήλατα. Εγώ χαίρομαι ότι χαίρεται και ο πρόεδρος του Συμβουλίου αλλά και η αρμόδια επίτροπος έχει εκφράσει την ικανοποίησή της ότι πρώτη φορά που ήρθε στο Κοινοβούλιο ήρθε με το ποδήλατό της. Αυτό ήταν ένα ιστορικό γεγονός ότι ουσιαστικά και τα τρία θεσμικά όργανα υποστηρίζουν το ε, ποδήλατο και όταν πήγαμε από το Λουξεμβούργο για να φάμε από το Συμβούλιο, πήγαμε με το ποδήλατο. Και ίσως και άλλοι υπουργοί το έχουν πράξει αυτό. Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να τα ακούσουμε. δημ. ακούς. Για τα θέματα επικουρικότητος και φυσικά έχει σημασία η επικουρικότητα. Η αστική κινητικότητα πάντα αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Λένε όλοι, α, αυτό είναι θέμα επικουρικότητας και οι πόλεις θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν μπορούν από μια μεριά να παίρνουν ευρωπαϊκά χρήματα και μετά σε επίπεδο εφαρμογή ακολουθούν στόχου αντίθετου από αυτού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν παίρνουν ευρωπαϊκά χρήματα, τότε πρέπει να αναλαμβάνουν και υποχρέωση εναντί τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματοποιούν ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε χρήματα και να λέμε όχι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την επικουρικότητα. Και αν θέλουμε να πετύχουμε στόχους ε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και να έχουμε μια ταχεία και αποτελεσματική κίνηση στις πόλεις, τότε θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση. Όπως είπε ο Γερμανός υπουργό η Υπουργός, ότι θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος της κίνησης που γίνεται προς τις πόλεις να αντικατασταθεί από τα εμπορικά τρένα και ελπίζω ότι μπορούν αυτά να επιτευχθούν. και το θέμα της παραγωγής χάλιβος επίσης. Αλλά για την ε, δημιουργία, για την παραγωγή ποδηλάτων υπάρχει, υπάρχουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ό,τι στη χαλιβουργία. Μόνο αυτήν την διάσταση να σκεφτείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την απασχόληση και για το μέλλον, το οικονομικό μας. Ξέρω ότι ο Φρανσό Μπάους έχει ε, αγωνιστεί για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα για τους σιδηροδρόμους και τα λιμάνια που συζητάμε χωρίς να προχωρούμε. Είναι παράξενο, είναι απίστευτο ότι ένας ευρωπαϊκός τομέας δεν επιτρέπει να υπάρχει πρόοδος στα θέματα αυτά για τους σιδηροδρόμους γιατί η Eurostat αρνείται να συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Συνδροδομικό Φορέα και να έχει τις απαραίτητες στατιστικές. Τότε είναι θέμα της Κομισιόν. Μιλάμε συνέχεια για, τα, για το μπλοκάρισμα από την πλευρά του Συμβουλίου, αλλά εδώ πρόκειται για την Κομισιόν. Τώρα, αναφερθήκατε στο ανταγωνισμό στην αεροπλοεία και εσείς και κύριε Φανχάγεν. Είναι βεβαίως μια μεγάλη δυσκολία γιατί υπάρχουν περιοχές όπως είναι τα κράτη του Περσικού κόλπου ή η Τουρκία όπου κάποιες αεροπορικές εταιρείες υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν το ίδιο ε, κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο εσείς θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις χώρες του Περσικού κόλπου και να πείτε αν θέλετε να έχετε συνεργασία πρέπει να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό. Θα πρέπει να σταματήσετε τι κρατικέ επιδοτήσει. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώ η Ολλανδική Προεδρία θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Και, θα... και η συνάντηση που έγινε στο Άμστερνταμ ήταν πολύ θετική για τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε τι προσπάθειε Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει ανταγωνισμό αλλά μόνο για ορισμένου. Το τελευταίο σημείο το οποίο ανέφερε η Γκεζίνε Μάισνερ. Άμα κοιτάξουμε το συνδεδομικό δίκτυο της Ευρώπης είναι ένα είδος κουρελού. Είναι ένα εμβαλωματικό σύστημα που επί 300 χρόνια έχουν αναπτυχθεί με, 200 τρο... με... με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα συστήματα. Δεν πρόκειται να είναι κάτι το οποίο θα κοστίσει πάρα πολύ να έχουμε μια ενοποίηση για ορισμένα θέματα και με ποιο τρόπο εσείς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε να υπάρξει στον τεχνικό τομέα μια σειρά από προτεραιότητες, να υπάρξει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα και τα κράτη-μέλη που παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια για τα εθνικά του σχέδια να προωθούν αυτήν την ενιαία προσέγγιση. Επίσης λοιπόν θέλω να τονίσω ότι για το τέταρτο πακέτο πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, ελπίζω θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία. Πέτε Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω του υπουργού που ήρθαν να μα απευθύνουν το λόγο. Νομίζω ότι τα περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη τεθεί από του συναδέλφου μου. Ήθελα μόνο να θίξω ένα ζήτημα και να το απευθύνω ω ερώτημα προ ε, την Ολλανδέζα Υπουργό. Εδώ και χρόνια Είστε γνωστοί για το ενδιαφέρον και την έμφαση που δίνετε στην τομέα των μεταφορών στη χώρα σας. Ε, όλες οι μορφές μεταφορών. Είστε ένα έθνος μεταφορών. Στη χώρα μου, τη Σουηδία, είχαμε κάποια μικρά ζητήματα ε, σε ό,τι αφορά το καμποτάζ και έχουμε μία σειρά τοπικών επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν ε, να κλείσουν εξαιτία του αθέμητου ανταγωνισμού. Ενώ ξέρουμε ότι σα έχετε ενισχύσει την νομοθεσία σα σε αυτό το τομέα. Πολλά μπορούν να γίνουν και στη χώρα μου, δυστυχώ δεν έχουμε κάνει αρκετά. Όμω υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτό το θέμα του καπατάζ. Ο νομοθέτης ε, δεν είχε εξετάσει όλε τι στοιχείε του ζητήματο. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιον ε, που έχει τις... Ε, σε μια συγκεκριμένη γέφυρα, για παράδειγμα, μπορεί ε, να έχουμε τελικά περιπτώσεις όπου κάποιος χωρίς να το θέλει να είναι παράνομος, γιατί περνάει απλώς μια γέφυρα από την μία πλευρά στην άλλη, από τη Σουηδία στη Δανία. Ακούσαμε και τους συναδέλφους. Σε ό,τι αφορά αυτή τη γέφυρα του Eurosund, εγώ πήγα εκεί, είδα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δείχνεις απλώς το διαβατήριό σου, πέντε δευτερόλεπτα και φεύγεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να διασύσει κανείς τη γέφυρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, η κινδυνολογία. Και πάλι όμως επανέρχομαι στην ομοθεσία για το καποτάζ που δημιούργησε το τέτοιο προβληματισμό σε ό,τι αφορά το κοινωνικό dumping που είναι άμεση απόρρια ε, αυτών των ε, κανονιστικών ρυθμίσεων. Ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα προς ε, την εκπρόσωπο των κάτω χωρών, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και εσείς είστε έθνος μεταφορών. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να διασφαλίσουμε αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Εντάξει, ακούσαμε τους συντονιστές και θα πρότεινα να απαντήσετε πρώτα και έχουμε άλλους 11 ε, οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Φρανσουά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ερτού, ο οποίος έθεσε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Μάλλον δύο από τον κύριο Ερτού και την κυρία Κίλενεν πήρα τα δύο αυτά τα ερωτήματα τα οποία ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσω να ομαδοποιήσω και να απαντήσω και τα δύο ερώτηματα. Ποια είναι η προσωπική μου άποψη σε σχέση με το τέταρτο σιδηροδομικό πακέτο και για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις ε, ε, δυσκολίες, ποια είναι η κληρονομιά που θα δώσουμε ουσιαστικά στην Ολλανδική Προεδρία. Για μένα το σημαντικό είναι μέχρι το Μάρτιο ή Απρίλιο να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το πακέτο στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Έχουμε επεξεργαστεί μια συμβαστική λύση ως Λουξεμβούργο και φυσικά εκεί κατευθυνθήκαμε σε μεγάλο βαθμό ακολουθώντας την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ακολουθώντας λοιπόν και την φιλοσοφία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό έδειξε και ο Τρίλογος όπου ήταν πολύ θετική η ατμόσφαιρα και γι' αυτό το λόγο εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι δυσκολίε τώρα είναι κυρίως όταν θέλουμε να, να αποκλίνουμε από αυτήν την ε, θέση και τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να αποκλίνω από αυτή τη φιλοσοφία που έχει υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ νομίζω ότι είναι λανθασμένο να κάνουμε νομοθετικά κείμενα τα οποία βασίζονται στη λογική ότι η Ευρώπη είναι ομοιόμορφη, ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ περιφερειών, ότι δεν υπάρχουν περιφερειακές ιδιαιτερότητες. και δεν μπορούμε να τα δούμε τα θέματα εξάλλου και μονάχα με μια εθνική και μονολογική. Αυτό θα μας οδηγήσει σε λανθασμένη αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι η συμβαστική λύση που επετεύθηκε, η οποία υποστηρίχθηκε και από την Κομισιόν και η οποία χάρηκε για την συμβαστική πρόταση του Λουξεμβούργου, ελπίζω ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία και όχι με διάφορα τεχνάσματα να γίνει μια προσπάθεια να ανατραπεί αυτό το οποίο επετεύχθη τον Οκτώβριο. Αυτό θα είναι σημαντικό για το σύνολο του πακέτου για τα συνδρομικά θέματα. Εξακολουθώ όμως να είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την τελική συμφωνία. Επίσης πιστεύω ότι η μέθοδος που ακολουθήσαμε και η μέθοδος του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι και ένα δίδαγμα για άλλους τομείς, θα είναι ένα υπόδειγμα για άλλους τομείς. Χάρηκα λοιπόν που επιτέθηκαν όλα αυτά, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι <clears throat> αυτή η μέθοδος μπορεί να μεταλαμβαδευτεί και σε άλλους τομείς διαπραγματεύσεων. Θέλω επίσης να πω ότι για τον πρώτο πυλώνα, για τον τεχνικό πυλώνα, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το να κλείσουμε αυτόν τον πυλώνα, τις διαπραγματεύσεις αυτόν τον πυλώνα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα έχουμε μία συμφωνία, από τη στιγμή που υπήρξε η συμφωνία για τον τρίτο πυλώνα στο Συμβούλιο, θα πρέπει να δώσουμε την θέση μας στο Κοινοβούλιο του ταχύτερο δυνατό και το κάνουμε. Στις 18 Δεκεμβρίου είχαμε τη γνωμοδότηση της Κομισιόν, ρωτήσαμε την Κομισιόν για τη θέση της, μας ε, παρουσίασε κάποιες μικρές δυσκολίες, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν ώστε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο να μπορέσει να εγκρίνει τα θέματα που συνάπτονται με τον τεχνικό πυλώνα. Δεν βλέπω να υπάρχει λοιπόν κανένα λόγο περαιτέρω καθυστέρηση. Είμαστε όλοι πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούμε να κλείσουμε το πακέτο και δεν πρέπει για αυτό το λόγο να αναβάλουμε καθόλου την ένδυση του τεχνικού πυλώνα. Αν λοιπόν εξακολουθήσουμε στην πορεία αυτή που ανέφερα σε σχέση με το τέταρτο πακέτο, αυτά δηλαδή τα οποία τη φιλοσοφία, τη γενική αντιμετώπιση που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω ότι στους επερχόμενους τριλόγους μπορούμε να προχωρήσουμε και στη συνέχεια το Μάρτιο να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν το παρακολούθησε αυτό. Έχουμε δει την αντίδραση της Κομισιόν. Νομίζω ότι το πρόσωπό σας τα, τα δείχνει όλα. Ισμαήλ, ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Στην προηγούμενη ερώτησή μου ίσως δεν είχα ε, αναφερθεί σωστά. Ε, ανέφερα κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν την Κομισιόν και όχι το Συμβούλιο. Ναι, ναι, ήταν πολύ σαφέ. Είναι πάρα πολύ καλό να μπορέσει η Κομισιόν να μας, εξασ, να ε, εκφράσει τη δική τη άποψη. Ναι, τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά, λέει ο πρόεδρο. Τώρα η υπουργό των Κάτω Συγγνώμη, η Ολλανδή, η κατοχωρήτησα υπουργό Βιμ. Δεν το είπα σωστά. Um, <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω την πρώτη ερώτηση στα Ολλανδικά, γιατί ήταν ε, ερώτηση του κυρίου Βαντερκάμπ. Νομίζω ότι ο κύριος Βαντερκάμπ με ρώτησε, ε, μου ζήτησε μάλλον ένα σχόλιο μεταξύ άλλων και για το θέμα των εκπομπών. Αυτή τη στιγμή αναπόκειται στο Κοινοβούλιο ε, να ψηφίσει μία πρόταση. Επομένω, ε, το μπαλάκι έχει πέσει στο δικό σα ε, γήπεδο αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα τι μορφή θα πάρουν τα άλλα δύο ζητήματα, για να αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο, τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση ε, για τα θέματα αυτά. Από ό,τι ξέρω λοιπόν ε, και το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται μία πρόταση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε και να πράγουμε και εκεί το διάλογο. Τρία συμβούλια βεβαίως ε, ασχολούνται με αυτό το θέμα και μεταφορών αλλά και περιβάλλοντος. Όλα αυτά βεβαίως υπό μία προεδρία, επομένως θα υπάρξει και μια συνεργασία, εννοείται. Τώρα, ε, για τις μικρές πλωτές οδούς, όπως αναφέρατε, και τη χρηματοδότησή τους. Η φιλοδοξία είναι πραγματικά και η αστική ναυσεπλοεία να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα και του ευρύτερου συστήματος μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και χρηματοδότηση της, για τη διαχείριση ε, και ε, συντήρηση και των μικρών πλωτών οδών ε, θα προσπαθήσουμε και μέσα στο 2016 να θέσουμε επιτάπητο στο ζήτημα αυτό για να είναι σαφές ότι είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί. Τώρα, να περάσω στα ερωτήματα του κυρίου Ερτούκ για το TTIP. Μεταφορές, ιδίως ε, οι θαλάσσιες μεταφορές, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσει για την TTIP, οι οποίες ακόμα λαμβάνουν χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν ακόμα να ε, προδικάσουμε τις συνέπειες της TTIP για τον τομέα των μεταφορών, Όμως ε, εν γέννη γιατί συζητήσατε την προσωπική μου γνώμη, αλλά αυτό καλύτερα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα είμαι εδώ με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Συμβουλίου, αλλά θεωρώ ότι μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα έχει ευνοϊκές προεκτάσεις, ανοίγοντας τα σύνορα και νέε αγορέ, μάλλον και για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Στην προσωπική μου γνώμη να μου τη ζητήσετε καλύτερα κάποια άλλη στιγμή. Μετά, με ρωτήσατε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες ε, της Ολλανδικής Προεδρίας ε, για τον φάκελο των οδικών μεταφορών. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες προτάσεις επί δικής μας Προεδρίας, ούτε προβλέπεται νομοθετική πρόταση. Ξέρουμε βεβαίως ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται ένα αντίστοιχο πακέτο και θα το παρουσιάσει νομίζουμε στο δεύτερο εξάμεινο του 2016 μετά την Ολλανδική Προεδρία. Εξετάσαμε τις κοινωνικές διαστάσεις κατά την προηγούμενη Προεδρία υπό τον κύριο Μπάους. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συζήτηση εκεί και το πιο σημαντικό σχόλιο από τα περισσότερα κρατημέλη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει ε, νέο κανονιστικό πλαίσιο, νέα νομοθεσία, αλλά καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού που ήδη έχουμε στην κοινωνική, σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση. Αυτό συνδέεται και με τα όσα αναφέρθηκαν για τους ΙΔΙΑ, γιατί πολλές χώρες εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τους κανόνες ε, επί των κοινωνικών διαστάσεων. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Νομίζω ότι η Κομισιόν θέλει να θίξει το ζήτημα των, της κοινωνικής διάστασης ε, του οδικού πακέτου. Δεν ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η πρότασή τους, αλλά μπορείτε ίσως να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς να δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Ο κύριος Έρτουκ επίσης ε, με ρώτησε και ο κύριος Βαντεκάμπ ε, και άλλα μέλη της Επιτροπής μας επένεσαν επειδή θέσαμε το ζήτημα των συνδεδεμένων ε, και αυτόνομων οχημάτων. Και με ρωτήσατε τι προτίθεμαι να κάνω μέσα στις επόμενες συνεδριάσεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά θετικά να αποκομίσουμε από την προώθηση της ε, εφιούς και πράσινης κινητικότητας, ιδίως και των αυτόνομων οχημάτων. Και από την πρωτολογία μου ε, είδατε ότι για μένα είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε χαμηλότερη καταναλώση καυσίμων, λιγότερα τροχαία ατυχήματα, ε, καλύτερη αξιοποίηση του, των δικών δικτύων και ζητήσαμε και από την Επιτροπή να το εξετάσει, όπως είπατε, θέλουμε να επιτύχουμε συμφωνία με όλα τα κράτη-μέλη και να το αποκαλέσουμε δήλωση του Άμστερνταμ για να δούμε τι πρέπει να γίνει ε, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου ή και απλοποίηση αυτού ε, και να δούμε επιμέρους στοιχεία πώς είναι ε, η προστασία του, της ιδιωτικής σφαίρας ζωής ή τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά για παράδειγμα στη συνδίκη της Βιέννας λέμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε τα χέρια στο τιμόνι. Και αυτό είναι αρκετά παροχημένο ε, σαν σκέψη, αν δείτε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τροποποιήσεις και θέλω να υπάρχει στήριξη όλων των κρατών μελών. Σημαντικό είναι να γίνει με ομοιόμορφο τρόπο. Βλέπετε, ας πούμε, στα τρένα ότι κάποιος ε, πρέπει ε, όταν, αλλάζει, όταν περνάει τα σύνορα πρέπει να αλλάξει και τι ε, προδιαγραφέ ασφαλείας του. Δεν θέλουμε να συμβεί το ίδιο σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Ζήλε τώρα και κυρία Μάισεν επίσης ε, έθεσαν κάποια ερωτήματα για τον κανονισμό υπηρεσιών στους λιμένες. Η γενική προσέγγιση που από το Συμβούλιο 2014 τηρεί τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν, ταυτόχρονα όμως εισάγει και στη μεγαλύτερη ευελιξία και περιορίζει το διοικητικό άκθος. Δεν ήταν εύκολο να επιτύχουμε συμφωνία ε, στο Συμβούλιο, όμως τον Οκτώβριο του 2014 καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί ενός ε, συμβαστικού κειμένου με ευρεία συνένεση. Το Συμβούλιο ακολουθεί μία δίκαιη, ρεαλιστική και ε, πρακτική προσέγγιση και θα ξεκινήσουμε, θα, μάλλον θα αποτελέσει βάση συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και για το μέλλον με το Κοινοβούλιο. Θέλω να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει. Δυστυχώ ε, δεν υπερψηφίστηκε σήμερα. Ε, και σα καλώ να υιοθετήσετε μία εντολή διαπραγμάτευση το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριο Ζήλια, επίση, ρώτησε ποιε είναι οι προθέσει μα σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό πακέτο και ιδίω τον πυλώνα ε, τη αγορά. Και ο κύριο Μπάου, νομίζω, πολύ εύγλωτα ανέφερε ότι είναι ένα συμβιβασμό μεταξύ πολλών χωρών. Μπορεί κάποιος να πει λοιπόν ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το συμβιβασμό, αλλά όταν επετέχθη ο συμβιβασμός όλοι χαρήκαμε που υπήρξε κάποιος συμβιβασμός. Είναι δύσκολο λοιπόν γιατί υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις, ακόμα και στο κοινοβούλιο οι απόψεις δίστανται. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σε βάθος συζήτηση για το τι είναι εφικτό και τι όχι. Πραγματικά ελπίζω να καταφέρουμε να επιτύχουμε συμφωνία μέχρι το Πάσχα. Η κυρία Μάισνερ. Α, κύριος Ήλε και πάλι ρώτησε για τη μετανάστευση. Ήδη έχω θίξει αρκετές φορές ε, αυτό το ζήτημα σε επίπεδο επιτροπή. Τώρα με ρωτήσατε ποια προβλήματα εντοπίζω σε ό,τι αφορά την μετανάστευση και την ε, σύνδεση του ζητήματος αυτού με το τομέα των μεταφορών. Το έχω δείξει πολλές φορές σε επίπεδο Δεν είναι στο θεματολόγιο ε, του, του Συμβουλίου Μεταφορών, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα και πάντα θα πρέπει να το έχουμε κατά νου γιατί ό,τι προκύπτει από ένα ε, Συμβούλιο Υπουργών επηρεάζει και άλλα Συμβούλια Υπουργών. Αυτό είναι σαφές. Ε, δεν αφορά δηλαδή μόνο τη μετανάστευση, αλλά και άλλους τομείς. Η κυρία Μάισνερ με ρώτησε πώς μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε ε, την πρόταση για την αεροπλοεία. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι το κάναμε ή θα το κάνουμε. Κανείς δεν ξέρει αλλά ξέρετε ότι είναι ένα ζήτημα δύο κρατών μελών. Ε, πρέπει να λυθεί το ζήτημα του Γιβραλτάρ. Η Προεδρία είναι κατεθειμένη να βοηθήσει όπου μπορεί. Δεν έχουμε επίσημο ρόλο να διδραματίσουμε, όπω ξέρετε. Είναι ζήτημα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και υπουργών εξωτερικών. Αν βρεθεί όμω λύση και αν μπορούμε εμεί να συμβάλλουμε. Βεβαίω και θα το πράξουμε. Και βεβαίως και είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε αυτούς τους φακέλους, όπως είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και τα δικαιώματα των, επιβατών. Κατανοώ ότι υπάρχει ισχυρότατη πίεση. Αν έχετε κάποια καλή ιδέα για να ξεμπλοκάρει ε, αυτή η υπόθεση, να μου την πείτε. Τώρα, είπατε σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και σε σχέση με ε, τον διεθνή τομέα της αεροπλοείας. Δεν ήταν σαφή η θέση τους ε, σε ό,τι αφορά μια νέα πρόταση για το κλίμα. Η ε, Συμφωνία των Παρισίων είναι σαφής για την ευθύνη και των δύο τομέων και η αεροπλοεία δηλαδή θα πρέπει να εισαγάγει μέτρα για να περιορίσει σημαντικά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Και είναι δική μα ευθύνη να εξακολουθήσουμε να τονίζουμε και από δική μα ε, πλευρά ε, αυτά τα στοιχεία, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική και θα διατηρηθεί αυτή η δυναμική στην ε, διεθνή αεροπλοεία. Πρέπει βεβαίω να εξετάσουμε και τι άλλε μορφές μεταφορών. Για τα ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων είναι σημαντικό τμήμα και στοιχείο και αυτό. Σημαντικό στόχο αν θέλουμε, οι δημόσιες συγκοινωνίε να γίνουν πιο ελκυστικέ. Όμως, τώρα αυτό πρέπει να γίνει μέσω κανονισμού. Μήπως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, ρύθμι, απαιτεί μάλλον ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχουμε και πολλές ε, επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και ίσως και η αγορά να μπορεί να το αναλάβει. Κύριος Κρέμερ. Μίλησατε για τα στατιστικά σε ό,τι αφορά τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Ξέρω ότι είστε υπέρμαχος ε, των σιδηροδρόμων κάποιος ανέφερε ότι είστε και υπέρ και των ε, αυτόνομων οχημάτων, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με τους σιδηροδρόμους. Η Ολλανδική Προεδρία ε, θέλει να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το φάκελο που έχει βρεθεί σε διέξοδο από το Δεκέμβριο του 2014 και πρέπει να αναθεωρηθεί το 8α που καλεί τα κράτη-μέλη να διεξαγάγουν μελέτες ε, για συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Το Συμβούλιο ζητά από το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε επιπλέον στοιχεία, ιδίως ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Όμως θεωρούμε ότι τα περισσότερα αιτήματα του Κοινοβουλίου ήδη καλύπτονται και από την DG Move και από άλλες ε, και με άλλες μεθόδους και νομικές πράξεις συμφωνήσαμε επί μια μη νομοθετική ε, λύσης με τη συμπερίληψη δεδομένων που ζητά το Κοινοβούλιο σε ένα μνημόνιο κατανόηση ε, μεταξύ Eurostat και DG Move. Η Κομισιόν όμως των πρόγραμμα εργασιών της 2016 ανέφερε ότι είναι διατεθειμένη να αποσύρει την πρόταση εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Ε, η κυρία Κρέμερ ζήτησε και για τις εντολές για τα κράτη του Περσικού του Περσικού κόλπου και πιο συγκεκριμένα για τον αθέμητο ανταγωνισμό και επίσης ε, ρώτησε περί ανταγωνισμού στην αεροπλοεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό στους σιδηροδρόμους και εντός ε, του τομέα της αεροπορίας Πιστεύω ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις μπορούν να, να βοηθήσουν σε τέτοια ζητήματα και ζητήματα περιβαλλοντικά και άλλα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Ε, πιστεύω ότι και η κανονιστική σύγκληση για θέματα όπως η ασφάλεια, ο έλεγχος των αεροπορικών εταιριών ε, μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο πιο ε, αποτελεσματικής διαπραγματεύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εστίαση λοιπόν στο θεμητό ανταγωνισμό θα αποτελέσει κομμάτι των στόχων μας. Κύριε Λεντγκρεν, με ρωτήσατε για την Ολλανδική νομοθεσία. Αλλά όπως σας είπα εγώ δεν βρίσκομαι εδώ ως Ολλανδή υπουργό, αλλά ως πρόεδρος όλων των υπουργών μεταφορών. Ε, με ρώτησε λοιπόν για την νομοθεσία περί καμποτάζ χρησιμοποιώντα τη γέφυρα Έρωσεντ ως παράδειγμα για το πόσο εύκολα τι εύκολο που είναι να αποφευθεί νομοθεσία για όλο αυτό. Το συζητήσαμε αυτό συζητώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο του πακέτου για τις οδικές μεταφορές το ερώτημα είναι πρώτα, αφορά την εφαρμογή. Κατά πόσο εφαρμόζουμε όλα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο στις διάφορες χώρες, πώς τα ελέγχουμε. Ε, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα του καμποτάζ και αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι το πρόβλημα έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με τη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και μετά πρέπει να δούμε κατά πόσο εφόσον έχει εφαρμοστεί παντού το, ο σχετικός κανονισμός πώς ρυθμίζουμε εκ νέου λεπτομέρειες. Ευχαρίστως να ακούσουμε τις ιδέες σας αν υπάρχουν και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη για περαιτέρω συζητήσει. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα όλες τις ερωτήσεις των μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα μισή ώρα. Έχουν ζητήσει 10 ακόμα βουλευτές ε, το λόγο. 1,5 λεπτό ο καθένας, σύντομα και συνοπτικά και μετά θα δώσουμε στους υπουργού τη δυνατότητα απάντησης και θα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση μετά από όλα αυτά. Ο Τζορτς Μπαχ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τις ευχές μου καταρχήν, τα συγχαρητήρια μου καταρχήν στον Πρόεδρο του στον Υπουργό του Λουξεμβούργου και τους συνεργάτες, τον κύριο Μπάους, νομίζω ότι έχουν κάνει πολύ καλή εργασία. Ε, είσαι Λουξεμβουργιάς, του τώρα ο πρόεδρος. Όχι. Μα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα του Κέσσαρ στο Κέσσαρι. Αν κάτι έχει γίνει καλά πρέπει να το πούμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για τις σαφείς δηλώσεις του σε σχέση με το συνδεδομικό πακέτο. Και εμείς φοβόμαστε ότι υπάρχει μια προσπάθεια τώρα να να ξυλωθεί το pullover κατά κάποιο τρόπο και από την πίσω πόρτα να δημιουργηθούν νέες ε, συνθήκες και να αλλάξουν οι συμφωνίες. Έχουμε λοιπόν αυτές, αυτούς τους φόβους και εμείς γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που έχει επιτύχει η Προεδρία του Λουξεμβούργου μαζί με τους Ολλανδούς συναδέρφους να συνεχίσουν να ακολουθούν τη σωστή γραμμή. Κύριε Υπουργέ Μπάους, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έχει γίνει με το θέμα της μέτρησης των τιμών των καυσαερίων στην ε, επιτροπολογία. Εμείς νιώθουμε απογοητευμένοι γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξες οι προσπάθειες που έχουν γίνει και με τις νέες εξελίξεις που προήλθανε θα ήθελα να θέσω το ερώτημα πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και για τον τομέα του κοινωνικού ντάμπινγκ θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εμπορευματική μεταφορά στον οδικό χώρο γιατί είναι φανερό ότι υπάρχει εκεί κάποιο dumping. Και περνάω αμέσω στην Ολλανδή Υπουργό. Σα ευχαριστώ και εσά πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Πώ βλέπετε λοιπόν και εσεί την εξέλιξη στα θέματα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μα το κοινωνικό dumping. Δεν θα ήθελα λοιπόν μετά από τη Λουξεμβουργική Προεδρία να προχωρήσουμε χωρίς καμία πρόοδο. Κάτι ακόμα και για τα δικαιώματα των επιβατών και τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ε, εθέρες και για το ΕΦΣΥ, το πρόγραμμα επενδύσεων του Ιούκερ, το οποίο όμως δεν αναφέρθηκε καθόλου σήμερα και παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τις επενδύσεις. Πού βλέπετε να υπάρξουν περαιτέρω πρόοδοι. Συγγνώμη που βλεπετε να υπαρξουν περαιτερω προοδες συγγνωμη που μακρηγορησα Ε, δεν σε διέκοψα. Η Λούση Άντερσον. Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που σας ε, βλέπω εδώ Αναφέρομαι κυρίως στο έργο σας και των δύο χωρών. Αναφέρομαι στην ε, δέσμευσή σας για περιβαλλοντικά φιλικές μεταφορές και εύχομαι όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι προεδρίες ε, να έχουν την ίδια δέσμευση. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για το έργο σας ε, τον Απριλίο για τις έξυπνες πόλεις και την κινητικότητα. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλά μέλη της Επιτροπής αυτής και είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε το ολιστικό ψήφισμα που πέρασαν το Σεπτέμβριο για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να αναφέρω μια πτυχή που ελπίζω να εντάξετε στο έργο σας, την ε, κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση των αναπήρων. Διότι είναι σαφές ότι, παρότι βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την επικουρικότητα, εάν μια ισχυρή προεδρία και η Κομισιόν ε, δείξουν το δρόμο, δείξουν πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες μεταφορές χωρίς αποκλεισμούς ε, προσπελάσιμες εντός των πόλεων ειδικότερα θα μπορέσουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Και μια άλλη γρήγορη ερώτηση. Ξέρετε ότι πολλοί από εμά έχουμε υπογράψει μια γραπτή διακήρυξη για τους σοβαρούς τραυματισμούς ε, στους δρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σοβαρό πρόβλημα Πολλοί από εμάς προσπογράψαμε ε, αυτούς τους, τους στόχους. Ε, μπορείτε να πιέσετε λίγο την Κομισιόν να κάνει κάτι. Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι στόχοι πραγματικά βοηθούν. Πάνω από 200.000 τραυματισμοί οδηγούν ε, σε σοβαρά προβλήματα στις ζωές πολλών ανθρώπων. Αλλάζουν τη ζωή ανθρώπων στην Ευρώπη και Ελπίζω να εισακουστώ σήμερα. Παρακαλώ, υπογράψτε την γραπτή διακήρυξη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζάκη Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Λουξεμβουριανή η Προεδρία. Έκαναν καταπληκτικές, καταπληκτική δουλειά και συμφωνώ με αυτό που είπε, ότι προσπάθησαν να κάνουν λίγα σε, ε, για το χρόνο που είχαν, αλλά καλά. Ελπίζω να ακολουθήσει και η Ολλανδική Προεδρία. Δύο σχόλια για το πακέτο για την αεροπορία. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια για την ε, μη στρατιωτική χρήση των drones. Έχουμε βρει τεράστια υποστήριξη για την κατεύθυνση που θέλουμε να εθετήσουμε για το θέμα αυτό. Οπότε ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση αυτή που έχει διατυπώσει το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω, επειδή το αναφέρατε κι εσείς, ε, το ζήτημα του ανταγωνισμού. Η Dutch East India ήταν η πρώτη πολυεθνική το 1602 ε, στον κόσμο ως Βρετανοί εμείς ε, όπως και εσείς οι Ολλανδοί είμαστε ε, παγκόσμιοι έμποροι και πρέπει να προσέξουμε πολύ ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε δεν μπορούμε να καθορίσουμε επακριβώς πώς χρηματοδοτούνται οι αεροπορικές εταιρείε των τρίτων χωρών σίγουρα θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό αλλά όπως δεν έχει δικαίωμα ε, μια τρίτη χώρα να μας πει τι να κάνουμε με τις επιχειρήσεις μας εδώ, ούτε εμείς έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Οπότε θέλω να πω ας προσέχουμε. Μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα έρμπα στο Α380 και το Α350 που παράγουμε εμείς, ε, ε, οι μεγαλύτεροι αγοραστές τους είναι οι εταιρείε του Περσικού κόλπου. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση αλλά θα έλεγα να προσέχουμε πώς κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Προσδοκώ να συνεργαστώ μεταξύ σας και ελπίζω να είμαστε επικοδομητικοί στο έργο μας και σίγουρα θα έχετε την υποστήριξη του ECR. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Παβέλ Τελίτσκα. Ευχαριστώ. Ένα μικρό σχόλιο από πλευρά μου, να ξεκονομήσω και χρόνο. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάουσα για τι προσπάθειε ε, που κατέβαλε το Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια τη Προεδρία του. Πολλά έχουν υποθεί ήδη από αυτού και κυρία, ε, κυρία Υπουργέ, συγγνώμη, σα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ε, Δράτωμα από κάτι το οποίο αποτελεί κοινό στοιχείο, στοιχείο μεταξύ Τσέχων και Ολλανδών και αυτό είναι η ευθύτητα. Στον τριμερή διάλογο για τι δημόσιες προμήθειε. Ο Πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα μίλησε για το πώ μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε τη δυναμική τη ιστορική αγορά. Μέχρι τώρα όμω ε, η θέση του Συμβουλίου κινείται προς εντελώ διαφορετική κατεύθυνση. Ε, Μα δείξατε μια εικόνα λοιπόν με αυτό το διθέσιο ποδήλατο. Όμω, πρέπει να γίνει ένα ποδήλατο με πολλέ ε, θέσει και κατευθύνσει. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με ε, την απελευθέρωση της δυναμικής και των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς. Απλώς δίνει τη δυνατότητα ε, να δώσουμε σύμβαση σε οποιονδήποτε υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Πρέπει λοιπόν ε, να πω ότι για πολλούς από εμάς η κόκκινη γραμμή είναι ο δικαιούχος να είναι ο πελάτης. Γι' αυτό δεν περνάει αυτή τη στιγμή στην θέση του Συμβουλίου όχι ως προειδοποίηση, αλλά ως θέση που έχουμε πολύ εδώ. Και μέχρι τώρα είναι απογοητευτικά τα στοιχεία. Όμως ε, κάτι θα καταφέρουμε τελικά, όσο γίνεται πιο γρήγορα βεβαίως, αλλά πρέπει να υπάρχει και ποιότητα. Ευχαριστώ κυρία Καραμεντιλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συγχαρώ την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου. Πραγματικά μας δείξατε μία τρομερή ε, συνεργασία και με εμά τους βουλευτές και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γέννη και δείξατε πόσο άξιοι είστε αλλά και το επικαθηματικό σας πνεύμα. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για μια κάπως ιστορική πράξη στο πλαίσιο ε, της Επιτροπής Μεταφορών του Κοινοβουλίου. Πετύχατε να υπάρξει τουλάχιστον μια δήλωση για τα ποδήλατα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα ως εισηγήτρια και για την αστική και βιώσιμη ε, κινητικότητα με ενδιαφέρει ιδιαίτερο αυτό το ζήτημα και πρέπει να το σχολιάσω. Θεωρώ ότι δείξατε και επιδείξατε πολύ καλή ε, βούληση, σημαντική, τρομερή αφοσίωση και ελπίζω ότι και η Ολλανδική ε, κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Τώρα, σε ποιο τεχνικό επίπεδο, πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η αλλαγή σκητάλης μεταξύ της Προεδρίας του Λουξεμβούργου και των κατοχωρών. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ σημαντική πρόκληση και το λέω αυτό και ως εισηγήτρια για την βιώσιμη ε, κινητικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι δολοφονικές οι εκπομπές. Είδατε τι συμβαίνει ε, και με, τα, με τη Volkswagen, το, οποίο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σχέση με τα, όσα θα έρθουν. Ελπίζω λοιπόν, είπατε και εσείς ότι τον Απρίλιο θα γίνει ένα φόρουμ για την ε, αστική και βιώσιμη κινητικότητα. Εγώ όμως θα ήθελα πραγματικά να, ε, υπάρχουν, να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, γιατί μιλάμε για τη δημόσια υγεία των πολιτών μας. Δεν μπορούμε πλέον να παίζουμε με τη δημόσια υγεία θίξατε και μιλήσατε και εσείς για την COP21 και τα καλά της αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν και εσείς ε, να επικεντρωθείτε στα αποτελέσματά της ε, για τις μεταφορές ε, και για τις ναυτικές μεταφορές. Είχαμε μια ιστορική συμφωνία, δεν πρέπει να μείνουμε εδώ λοιπόν και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ανοίξει το ζήτημα, πραγματικά όμως να ανοίξει το ζήτημα και του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Κριστίνα Η Μαρή Κριστίνα Ρούτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μπάους, στο τέλος της Λουξεμβουργικής Προεδρίας είναι φανερό ότι υπήρξαν πολλές ε, δηλώσεις, πολλές δεσμεύσεις, αλλά λίγες πράξεις. Το ευρωπαϊκό σχέδιο που μας πουλάνε σε κάθε νέα προεδρία φαίνεται ότι είναι πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό γίνεται για απλού λόγου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τι προκλήσει της παγκοσμιοποίηση και βλέπουμε πόσο καθυστερούν ορισμένε διαπραγματεύσει και αυτό λόγω υπερβολικής ε, γραφειοκρατίας που δεν μπορούν να κατανοήσουν και οι πολίτες μας. Νομίζω ότι ο ρόλος της Προεδρίας του Συμβουλίου είναι να εφεύρει συγκεκριμένε λύσεις που μπορούν να αποσπάσουν τη συμφωνία των κρατών μελών. Κύριε Μπάους, ναι, από την Προεδρία σας είναι δύο πράγματα τα οποία έχουμε κρατήσει. Το ποδήλατο που μπορεί να είναι μια μελλοντική λύση για πολλά προβλήματα αφενός και αφετέρου το ότι η πολιτική μεταφορών θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τους στόχους της COP21. Εγώ μεγαλύδα. Ξέρετε ότι οι Γάλλοι αγαπούν ιδιαίτερα το ποδήλατο. Βλέπετε πόσο δημοφιλής είναι ο γύρο τη Γαλλία, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που του απασχολεί. Γι' αυτό θέλω να στραφώ σε εσά, κυρία Σούλτ Φανχάχεν. Η Ολλανδική Προεδρία θα πρέπει να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια να υπερασπιστεί τις εταιρείε τις που παράγουν αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα έναντι των διεθνών πιέσεων. Γιατί οι διεθνεί πιέσει μπορούν να καταστρέψουν αυτές τις βιομηχανίες προς όφελος των Ασιατών και Αμερικανών ανταγωνιστών τους. Θέλετε να έχετε ένα παγκόσμιο σύστημα για ποσοστώσεις εκπομπών από την αεροπορία. Μα οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν να υποστούν σοβαρούς και αυστηρούς ελέγχους, αντίθετα από ό,τι θα γίνεται σε πολλές τρίτες χώρες για την ε, ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το θέμα της ε, εισβολής των μεταναστών, στα, των μεταναστών στα πλοία και επίσης σε συνδεδομικούς σταθμούς όπως έγινε στο Καλέ πρόσφατα. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους ε, πολίτες μας το θεωρούν αυτό ότι είναι ένα αστείο. Αλλά ξέρετε ότι ο γαλλικός τύπος ανέφερε ότι θα υπάρξει μια, ότι εφαρμόστηκε μια απόφαση σε εσά στις, ε, στις, στις κατοχώρες σε σχέση με τους ε, ε, εκπαιδευτές οδηγών που ουσιαστικά παίρνουν το αντίτιμο των υπηρεσιών τους σε σεξουαλικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ναι, παρόλα αυτά πρέπει να σας διακόψω. Δεν μπορείτε έτσι όταν οι άλλοι να μιλάνε 1,5 λεπτό, εσείς να μιλάτε το διπλάσιο. Τους θέτετε σε μειονεκτική θέση. Σας έκανα δύο φορές νεύμα και εσείς δεν έχετε αντιδράσει. Περνάμε στην κυρία Λουγασένσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ξέρω ότι είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς ως Προεδρία όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη και φυσικά και πολλές οι προσδοκίες που τρέχουν οι Ευρωπαίοι από μια Προεδρία. αναλύσουμε λοιπόν τις ε, προεδρίες δεν μπορούμε ποτέ να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μία προεδρία έχει καταφέρει και να ξεκινήσει και να τελειώσει μια διαδικασία για ένα θέμα. Είναι τόσο πολύπλοκα τα θέματα αυτά που πάντα πρέπει να υπάρξει μια αλληλουχία προεδριών που θα το πετύχουν αυτό. Είναι τόσο πολλά τα πολιτικά θέματα που είναι απαραίτητα για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση για τα θέματα αυτά. αλλά θέλω και εγώ να επανέλθω στα προβλήματα τα οποία ανέφεραν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι οι μεταφορές σημαίνουν εκατομμύρια θέσεων ε, απασχόλησης. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός. Και τώρα θα ήθελα να ακούσω το εξής από τον κύριο Υπουργό. Μίλησατε για κοινωνικό ντάμπινγκ. Αλλά δεν πρόκειται για κοινωνικό ντάμπινγκ, πρόκειται για στρεβλώσει σε οικονομικό επίπεδο. Σε όλες τις ε, <clears throat> προτάσεις υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα κοινωνικά θέματα. Δεν πρέπει όμως να πάρουμε μέτρα τα οποία θα εμποδίσουν τη διατήρηση των ε, θέσεων εργασίας και θα εμποδίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εταιρεών. Πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας. Φαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία για το έργο της και ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας ε, δίπλα στην Ολλανδική Προεδρία. Δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο οπότε θα επικεντρωθώ μόνο στην Ολλανδική Προεδρία και θα συνεχίσω στα Ολλανδικά μου το επιτρέπετε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την πολύ επιτυχημένη αυτή συνοδογραφία για την αεροπλοεία. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ε, και μια πολύ καλή αρχή για μια επιτυχημένη Ολλανδική Προεδρία. Ένα ερώτημα να σας απευθύνω που αφορά την αεροπλοεία. Την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της ίδιας αυτής ε, συνόδου ε, για την αεροπλοεία ο διευθυντής της ΕΑΣΑ έκανε την εξή πρόταση που αφορούσε ακριβώς την πρόταση και την ιδέα να έχουμε μια, έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που θα ασχολείται ε, ε, με, το, με την ασφάλεια σε ό,τι αφορά την αεροπλοεία, ιδίως σε ό,τι ε, αφορά και περιοχές σύγκρουσης. Ποια είναι η δική σας στάση και θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει και αναθεώρηση ε, του βασικού κανονισμού για την ΕΑΣΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Άντρο a luxemburgi elnökség fél éve során a közlekedési ágazat szempontjából. Ευχαριστώ. Η Προεδρία έχει δώσει και στο παρελθόν θετικά αποτελέσματα στον τομέα των μεταφορών. Καταρχήν καταφέραμε να κλείσουμε να κλείσετε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το τεχνικό πυλώνα στο συνδρομικό πακέτο. Τώρα η ελπίδα μας είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει συγχρόνως να προωθήσει την συμφωνία για τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα, ακόμα και αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Μαρτίου που είπε ο κύριος Υπουργός. Θέλω επίση να ευχαριστήσω <clears throat> την Λουξεμβουργική Προεδρία για την αφοσίωση με την οποία έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά το προηγούμενο εξάμεινο και στους ε, τριλόγους. Η ελπίδα μας είναι ότι προτού περατωθεί η προεδρία των κάτω χωρών θα μπορέσουμε να κλείσουμε και τους υπόλοιπους πυλώνες στο πακετό συνδρομικών θεμάτων. Αυτό ήθελα να πω ως σκιώδης του ΕΛΚ για τα θέματα αυτά και επί Τροχάδιν, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές. Μιλήσαμε για την κοινωνική διάσταση και για μας στο ΕΛΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει σεβασμός των οδηγιών που έχουν να κάνουν την εσωτερική αγορά και έτσι να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ποια είναι η κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη υπάρχουν περιπτώσεις που ορισμένε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν πολύ χαμηλότερες αποδοχές και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Περιμένουμε από την Ολλανδική Προεδρία να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ε, συναφείς πτυχές. Θέλω να σας ευχηθώ λοιπόν κάθε επιτυχία, όχι μόνο για το συνδρομικό πακέτο, αλλά και για όλα αυτά τα θέματα. Μαρινέσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Λουξεμβουργική Προεδρία και την Ολλανδική Προεδρία. Η Κομισιόν έχει καταβάλει πολλές ε, προτάσεις ε, εντός του ΣΕΦ για επιμέρους έργα και στα τέλη του 2016 τα κράτη-μέλη είναι μάλλον υποχρεωμένα να παρουσιάσουν στρατηγικές για το στο πλαίσιο των συμφωνιών, αλλιώς δεν θα λάβουν κονδύλια. Επομένω, ε, σα ζητώ στο σχέδιο προπολογισμού 2017 να έχουμε αναπλήρωση των κονδυλίων για την ε, λειτουργία διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Ε, το Connecting Europe και να εγκριθεί ταυτόχρονα και η στρατηγική για τις μεταφορές για να έχουμε ακριβώς ε, το συντονισμό μεταξύ κρατών μελών. Για ολοκληρωθούν και ευρωπαϊκοί διάδρομοι. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα έργο στην Ανατολή, ένα στο Βορρά και ένα στο Νότο. Δεν είναι κάτι χρήσιμο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, η μοναδική λύση για το πακέτο αεροπλοείας θα είναι να αρχίσουμε να θέτουμε ζητήματα επιτάπητο και να γίνεται πραγματική συζήτηση. Ιδάλω δεν θα υπάρξει ποτέ επίλυση του ζητήματο. Εάν ξεκινήσει η συζήτηση, θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και τώρα δίνω το λόγο στους δύο υπουργούς για να μπορέσουν να απαντήσουν, αλλά παρακαλώ πέντε λεπτά ο καθένας. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί, το ερώτημα του κυρίου Μπαχ. Δυστυχώς, ε, κύριε Μπαχ, και πάλι θα πρέπει ε, να μιλήσω για τα ίδια και τα ίδια δεχομένω, ε, αυτή τη φορά για τα οχήματα. Η απάντηση είναι σαφή. Στην Επιτροπολογία έχουμε δύο χώρες που ε, έμειναν σταθερές μέχρι το τέλος, Λουξεμβούργο και κάτω χώρε για να έχουμε πιο αυστηρά πρότυπα. Όλες οι υπόλοιπε ήταν κατά. Προσωπικά λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πραγματικά να ε, αξιοποιήσει τη δύναμή του, την ισχύ του για να βελτιωθούν τα όσα αποφασίστηκαν μέσω επιτροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ, Μελανή Φούτφαν. Ελπίζω να τα καταφέρω εντός του πεντάλεπτου, γιατί πολλά έχουν ε, τεθεί. Θα μιλήσω λίγο πιο γρήγορα λοιπόν. Ο κύριος Μπάχ με ρώτησε για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν έχουμε ξεχάσει βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Ήδη το συζητήσαμε ε, και στην ε, συνάντηση της περσμένης εβδομάδας στη Χάγη, που ήταν ε, συζήτηση σε υψηλό επίπεδο για τις μεταφορές και περιμένουμε για την πρόταση της Κομισιόν μέσα στη χρονιά. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό σύστημα. Σε κάθε δυνατή ευκαιρία θα το συζητούμε. Μετά με ρωτήσατε για την εξελίξει ότι αφορά το ΕΦΣΥ σε σχέση με τις μεταφορές. Στην συντομία είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο γιατί παρέχει δυνατότητες και για τις υποδομές ε, πράσινης ενέργειας, καθαρής ενέργειας ε, συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, σε παραδοσιακά έργα υποδομών. Πρέπει λοιπόν τώρα να λάβουμε κάποιε αποφάσει και σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει για την ενδιάμεσα αναθεώρηση, όμω είναι σημαντικό να δούμε ε, τα επιμέρου μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην επόμενη περίοδο. κυρία η κυρία Άντσον και η κυρία Ντάλη ε, επεσήμαναν τη σημασία της πράσινης κινητικότητας. Έχουμε άτυπες ε, συναντήσεις και στο Συμβούλιο Μεταφορών και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα παράλληλα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή ποτέ. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να τα εξετάσουμε από κοινού αυτά τα ζητήματα και τα θέματα κινητικότητας και περιβάλλοντος. Και βέβαια η επικουρικότητα κάποιες φορές μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Είναι σημαντικό όμως να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, βέλτιση των πρακτικών και αυτός είναι σημαντικός ο ρόλος και της Ευρώπης σε αυτό το σημείο. Τώρα για τα τροχέα, τους τραυματισμούς, ακόμα και τους θανάτους. Όλα αυτά θα αποτελέσουν ε, τμήμα του πακέτου για τις οδικές μεταφορές. Και... Το συζητήσαμε στην περασμένη συνάντηση για τη διάρκεια μας Μαρινού ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη χώρα μου αυτό τα πάντα ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω όμως ότι θα, υπάρξει, θα συμπεριληφθεί στο πακέτο για τις οδικές μεταφορές. Μετά, Η κυρία Φώστερ με ρώτησε για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones, ε, που θα αποτελέσουν τμήμα των διαπραγματεύσεων για το πακέτο αεροπλοείας. Νομίζω λοιπόν ότι η δουλειά που έχετε κάνει θα ε, μας φανεί χρήσιμη και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και μας ε, ζητήσατε να προσέξουμε ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα. Γιατί όπως είπατε είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε ότι και οι τρίτες χώρες ε, θα λειτουργούν με διαφάνεια και δικαιοσύνη στις ε, δραστηριότητές τους. Βεβαίως ε, θα υπάρξει συζήτηση και από αυτού, πώς δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Κύριο Πάφελ, την Τλίτσκα, δεν με ρώτησε κάτι, έθεσε όμως ένα σχόλιο. Είναι σημαντικό ο πελάτης να είναι δικαιούχος κατά τις διαπραγματεύσεις για την αεροπλοεία. Και βεβαίως έχετε δίκιο. Νομίζω ότι ήδη απάντησα κάποια άλλα ερωτήματα. Μετά με ρωτήσατε για την εθνική αδειοδήγηση. Σε αυτό όμως είναι εθνικό ζήτημα. η κυρία Λουκασούφσκα. Ελπίζω να το λέω σωστά. Μου είπατε ότι είναι σημαντικό να δούμε και την άλλη πλευρά της ανταγωνιστικότητας. Να μην ρυθμίζουμε μόνο το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πάντα μιλούμε και για ε, δίκες, συνθήκες εργασίας οι θεμητές. Αυτό μπορούμε να το δούμε από την άλλη πλευρά του dumping. Ο κ. Βενίσελμπερκ με ρώτησε για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που θα είναι αρμόδιος για τις ε, ασφαλείς ε, αεροπορικές τροχές, οι γραμμές, οι ζώνες και θα το εξετάσουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού ΕΑΣΑ. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ξέρετε και μετά το ατύχημα με την MH17 είναι σημαντικό πλέον αυτό το ζήτημα, όχι μόνο για τις κάτω χώρες, αλλά και για άλλες ε, χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, στον κανονισμό ΕΑΣ θα το εξετάσουμε, αλλά εδώ δεν εκπροσωπώ μόνο τις ε, κάτω χώρε, αλλά όλους ε, τους υπουργούς μεταφορών. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Κάτι έχω ξεχάσει. Όχι. Εντάξει. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας προφανώς, για τις απαντήσεις που μας δώσατε για την πολύ καλή συμμετοχή που υπήρξε εδώ επίση και από τα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλω να ευχαριστήσω και για την πολύ καλή συζήτηση η οποία αφορούσε και το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έλευσή σας.